συγκεκριμένα το τι σημαίνει αυτό για το ηθικό ρίσκο των κρατών, τον ηθικό κίνδυνο των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. κύριος Μαριάν Μαρινέσκο από την Επιτροπή Έρευνας και ε, Βιομηχανίας.